Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντάκτες των ψηφισμάτων. Πρώτα ο συνάδελφος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι τόσο συχνό να ερχόμαστε εδώ και να χαιρόμαστε για τη λήξη ενός πολέμου, όπως ε, πραγματικά συνέβη το 2009 στη Σρι Λάγκα. Στη συνέχεια συστήθηκε το 2010 Επιτροπή Συμφιλίωσης και έχει αρχίσει και ε, στο μεταξύ η αποναρκοθέτηση. Τον Αύγουστο συστήθηκε μια ερευνητική επιτροπή για ε, τους αγνοουμένους και έγιναν στο μεταξύ στη Βόρεια Επαρχία εκλογές. Όλα αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Δυστυχώς υπάρχουν όμως και πάλι μαύρα σύννεφα στον ορίζοντα διότι ταυτόχρονα βλέπουμε να έρχονται συγκρούσεις, να γίνονται επιθέσεις σεξουαλικές, ε, απειλές γενικότερα να ε, εκτοξεύονται κατά της ε, δικαιοσύνης και συνολικά υπάρχουν και οι απροστάτευτες χείρες ε, πολέμου, οι οποίες υφίστανται ιδιαίτερες απειλές. Γι' αυτό η Σιλάνκα θα πρέπει αμέσως να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται μια επιτροπή που να εξασφαλίζει ότι εκείνοι που ε, έχουν ε, κάνει εγκλήματα πολέμου, εκατέρωθεν των αντιμαχωμένων πλευρών, να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη για να επέλθει και η τιμωρία τους κατατέθηκε μια έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη, πράγμα απαραίτητο, αλλιώς θα συστήσει ιδιαίτερη εξεταστική επιτροπή ΟΗΕ. Ε, θα πρέπει οι εκκληματίες πολέμου να λογοδοτούν πάντα ενώπιον των δικαστηρίων. Και όταν κάποιος έχει πέσει θύμα ε, βίας, είναι πιο εύκολο να ε, το ξεχάσει, να το συγχωρέσει και να συνεχίσει τη ζωή του όταν βλέπει τον θήτη του και τον δράστη να τιμωρείται. Ευχαριστώ πολύ κύριε.